Υπότιτλοι AUTHORWAVE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 Αρχίζουμε λοιπόν την ψηφοφορία, το πρώτο θέμα. Κυρία Ιντφελτ, διαδικαστικό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα συνάδελφοι, ακούσαμε την, ε, το χαιρετισμό του Προέδρου της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης. Πολύ σημαντικό γεγονός. Με αυτή την ευκαιρία έχω να κάνω μια παράκληση.